έκθεση Σφίντον όσον αφορά τις, τις δυνατότητες να επιβάλλει ε, κυρώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στατιστικές πληροφορίες που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έκθεση του κ. Γκουαλτιέρη. Ξεκινάμε με τους εισηγητές, τέσσερα λεπτά ο καθένας. Ο κ. Γκουαλτιέρη ξεκινάει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλήθη να τοποθετηθεί στη διαδικασία της διαβούλευσης στην πρόταση της αναθεώρησης που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο Συμβούλιο. Αφορά τον κανονισμό για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών. Είναι ένας κανονισμός που μαζί με αυτό που αφορά τις εξουσίες Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προβλέπει να επιβάλλει ε, κυρώσεις. Ε, είναι σημαντικό πλαίσιο της συλλογής στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πρόταση ε, δράζεται επί του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας που σε ισχύ και που δίνει νέες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δημιουργεί την αναγκαιότητα επικαιροποίηση των διαφόρων μηχανισμών συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων. Από τη στιγμή που εθετήθηκε η νομοθετική πράξη, από τη στιγμή που θα εθετηθεί, θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα να επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία με παρόμοιο τρόπο όπως κάνουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες που ασκούν ε, καθήκοντα ε, ε, εποπτείας για την χρηστή διαχείριση. Θα μπορεί επίσης να στοιχεία που συνήθως κάνουν οι εθνικοί φορείς εποπτείας για σταθερότητα του χρηματοστικού συστήματος και το ευρωπαϊκό σύστημα σταθερότητας στο αναγκαίο επίπεδο λεπτομέρειας για την επίτευξη των στόχων και στα πίσω των αρμοδιοτήτων. Στις 11 Νοεμβρίου ε, στην Επιτροπή ΕΚΟΝ ε, ενέκρινε την πρόταση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τάπεζας. Ε, συμπληρωμήθηκαν κάποιες προτάσεις για να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της εκθέσεως. Οι τροπολογίε που υπέβαλα ω εισηγητή έχουν σαν στόχο να εγγυηθούν πιο καλή διαβίβαση των στοιχείων και καλύτερη προστασία του εμπιστευτικού τους χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, μια τροπολογία προβλέπει την υποχρέωση για τις αρχές και τους φορείς που δέχονται τις πληροφορίες ε, εμπιστευτικές πληροφορίες, να υιοθετήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε να μπορούν να εγγυηθούν την προστασία των αλόγων δεδομένων. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ ενέκρινε και άλλες τροπολογίες που ενισχύουν κάποια σημεία που δεν καλύπτονται από τις συστάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα, ενισχύεται η διαφάνεια Όσον αφορά τη δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να δημοσιοποιεί τι αποφάσει τη που αφορά συγκεκριμένε κατηγορίε ε, ε, ε των διαφόρων πελατών και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ε, και αναφορές, σημαντικές αναφορές στην αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τον ορισμό και την επιβολή των υποχρεώσεων στατιστικής επισήμανσης και όσον αφορά τις κυρώσεις εισάγεται μια σαφής διάκριση μεταξύ αμέλειας και εκπροθέσεως παραβίασης σε περίπτωσης παραβιάσεως στη μεταβίβαση σε στοιχείων από τις υπηρεσίες μια πτυχή που αφορά κυρίως την, ε, στον σεβασμό της αρχής αναλογικότητας. Η οθέτηση αναθεώρησης έχει ιδιαίτερη σημασία συνεπώς διότι μπαίνει στο γενικότερο πλαίσιο αυξήσεως της εποπτικής εξουσίας ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Τραπεζικής Ένωσης. Θα ήθελα να δεχθεί ευνοϊκά ε, το Κοινοβούλιο τις προτάσεις της Επιτροπής ΕΚΟΝ και έτσι να επιτρέπει μια ταχεία έγκριση από πλευράς του Συμβουλίου και βεβαίως ε, υπήρξε και ευρεία συνένεση όσον αφορά την έκθεση και γι' αυτό ευχαριστώ τους κοιόδης συγκητέ και τις διάφορες πολιτικές ομάδες συνεργασία τους και δίνει αυτό άλλο ένα κίνητο στο Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Σουίνμπορν έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Χίλ, καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον ε, συντάκτη της αρχικής ε, έκθεσης. Εγώ θα προσπαθήσω να συνεχίσω στη βάση αυτή τη ε, έκθεση και τη δική του μεθοδολογία. Επίση, θα ήθελα να ευχαριστήσω του σκιώδει συγητές από όλε τι πολιτικέ ομάδε για τη συνεργασία του σε αυτή την έκθεση. Και παρά τι κάποιε διαφορέ, ε, ελπίζω ότι αυτή η θετική βολή θα επεκταθεί σε όλες τι εκθέσεις που θα ψηφιστούν αύριο. Στην τελευταία θητεία έγινε μια αλλαγή στο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντί να δρά σαν κεντρική τράπεζα με αρμοδιότητα επί της νομισματικής πολιτικής της δώσαμε την αρμοδιότητα να εποπτεύει τις μεγαλύτερες ε, τράπεζες στην Ευρωζώνη και με δυνατότητα για χώρες εκτός της Ευρωζώνης επίσης να συμμετάσχουν, να προσχωρήσουν σε αυτό το μηχανισμό η ΕΚΤ θα συνεχίσει βεβαίως να είναι ανεξάρτητη από πολιτικές επιδράσεις. Είναι επιτακτικό ότι στη νέα της λειτουργία ως εποπτικό όργανο να λογοδοτεί. Στο πλαίσιο των τριλόγων το Κοινοβούλιο προσπάθησε να εισάγει μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτές τις λειτουργίες της ΕΚΤ. Ε, δεν κάναμε τεράστια βήματα προς τα μπρος, ωστόσο υπάρχει ένα κομμάτι δημοκρατικής λογοδοσίας ε, και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση να αυξήσουμε την διαφάνεια. Στην, στο αρχικό σχέδιο έκθεση, όταν η ΕΚΤ επέβαλε κυρώσει σε ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό, μπορούσε να αποφασίσει κατά πόσο η απόφαση αυτή θα έπρεπε να κοινοποιηθεί και δεν προβλέπονταν καθόλου προθεσμίε. Ήταν εντό εντολή τη να το κοινοποιήσει ή όχι. Ωστόσο υπάρχουν αποχρόντες λόγοι ε, σε κάποιες ε, συγκυρίες να μην, ε, να μην δημοσιοποιούνται επιβολές κυρώσεων. Όταν για παράδειγμα μια, όταν υπάρχει κίνδυνος χρηματοπιστωτικής αποσταθεροποίησης το να είναι στο πρώτο φύλλο μιας εφημερίδας ε, δημιουργεί ένα κίνδυνο για ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό εξασφαλίσαμε μια προθεσμία τριών ετών, ούτως ώστε η ΕΚΤ ε, δεν θα πρέπει να ξεπεράσει αυτή την προθεσμία των τριών ετών για την, ε, όσον αφορά την κοινοποίηση της επιβολής κυρώσεων. Ε, εάν ε, θεωρήσουμε ότι οι κυρώσεις ε, συνεπάγονται στη λύτευση της φήμης ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού θεωρώ ότι είναι λογικό να επιτρέπεται μια, η παράταση αυτής της προθεσμίας και θα πρέπει να βασιζόμαστε μόνο σε ε, σοβαρές ε, καταγγελίες. Θα πρέπει να είναι έντιμη αυτή η διαδικασία αποκάλυψης των ε, τραπεζικών στοιχείων. Μόνο έτσι θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της ΕΚΤ και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο και οι πολιτικές ομάδες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την αύξηση της διαφάνειας αυτής της λειτουργίας. Ειδικά στην έκθεση Γκουαλτέρη έχω λίγα πράγματα να προσθέσω γιατί η ποιότητα του κανονισμού εξαρτάται από την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων ε, στους οποίους βασίζουν το έργο τους οι επόπτες. Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να έχουμε ποιοπτική εποπτεία είναι ποιοτικά στατιστικά στοιχεία. Γι' αυτό θα υποστηρίξω την έκθεση του κυρίου Γκουαλτιέρη στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ο Λόρδο Χίλ τώρα για την Κομισιόν για τρία λεπτά. Έχω ευγνωμονώ. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε τα συστατικά στοιχεία τη ΕΚΤ και τη κυρώσης που επιβάλλει ΕΚΤ και θέλω να συγχαρώ του δύο συγγητές για το έργο του η σύσταση των κυρώσεων τη ΕΚΤ είναι σημαντική γιατί είναι τμήμα της εφαρμογής Τραπεζικής Ένωσης και το χρειαζόμαστε γιατί θα δώσει στην ΕΚΤ τα μέσα να επιβάλλει την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Νομοθεσία και τις αποφάσεις της. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν υποστηρίζει πλήρως τους στόχους της ευθύς και καθώς οι κυρώσει μπορεί να έχουν ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο προς τη φήμη και οικονομικό αντίκτυπο θα πρέπει και μπορεί να υπάρχει και προσφυγή στα δικαστήριο, θα πρέπει να έχουμε σαφείς ε, κανόνες και ασφαλή δικαίου. Η Κομισιόν ε, δεν ανησυχεί με την προσέγγιση που έχει ακολουθήσει η ΕΚΤ στην σύσταση της υπηρεσίας. Η νομική υπηρεσία της Κομισιόν όμως ε, έχει εντοπίσει δύο προβλήματα της σύστασης και του κανονισμού για τον ενίο αποπτικό μηχανισμό. Ένα από αυτά τα σημεία σχετίζεται με ένα θέμα νομικής βάσης ε, και αφορά την εξουσία επιβολής ε, κυρώσεων, όχι μόνο ε, της των αποφάσεων της ΕΚΤ, αλλά και του άμεσου εφαρμοστέ νομική νομοθεσία και το άλλο αναφέρεται στην επιβολή κυρώσεων. Τώρα, το προ το προτείνει ε, τη δυνατότητα να καθυστερήσει η έκτετη δημοσίευση των κυρώσεων. Εγώ κατανοώ την λογική και βλέπω γιατί η ΕΚΤ μπορεί να θέλει αυτή τη διακριτική ευχέρεια. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα νομικό πρόβλημα, δεν ταιριάζει με τον κανονισμό ε, για τον νέο προοπτικό μηχανισμό που λέει ότι είτε υπάρχει προσφυγή ή όχι, θα πρέπει να υπάρχει δημοσίευση της κύρωσης από την ΕΚΤ. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα για τα επόμενα βήματα. Η Κομισιόν θα υιοθετήσει τη δική της γνωμοδότηση τις επόμενες εβδομάδες και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την ΕΚΤ για να έχει η ΕΚΤ όλα τα απαραίτητα μέσα για να εφαρμόσει την τραπεζική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία. Στι 13 Οκτωβρίου δημοσίευσε την ε, γνώμοδότηση της Κομισιόν. Ε, καλωσορίζουμε την ευθυγράμμιση ε, της συλλογή δεδομένων με τις νέες αρμοδιότητες της ΕΚΤ στον τομέα της προληπτικής εποπτείας. Θα μπορούν να στέλνονται νέες απόρριτες πληροφορίες σε όλες τις αρχές που είναι υπεύθυνε για τη μακροοικονομική εποπτεία. Επίσης, μειώνεται το άχθος για τις επιχειρήσεις, καθώς άπαξ πρέπει να συλλέγονται τα στοιχεία. Καλωσορίζουμε λοιπόν την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμφωνούμε με την άποψη που εκφράζεται στην έκθεση εικόν για το απόρριτο των στατιστικών πληροφοριών και είμαι ικανοποιημένα με όσα προτείνεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς τρία λεπτά. Συγχαρητήρια. Ο κύριος για δύο λεπτά για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως ΕΛΚ χαιρετίζουμε βεβαίως τη σημερινή συζήτηση, αλλά θα ήθελα καταρχήν να υπάρξει μια διευκρίνηση των αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ όσον αφορά τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων και των στατιστικών ε, στοιχείων. Γιατί η ΕΚΤ δεν μπορεί να δρά αυθαίρετα. Η ΕΚΟΝ ε, ήδη εξέφρασε την ε, θέση της και εμείς ε, οι βουλευτές θέλουμε ε, να ε, θα εκπληρώσουμε το καθήκον ελέγχου. Βεβαίως τα εμπιστευτικά δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά. Ως ΕΛΚ ωστόσο θα ήθελα να διατυπώσω κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά το, την εμβέλεια των στατιστικών στοιχείων. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει κάποια αναλογικότητα. Ε, και ε, δεν θα πρέπει να υπάρξει υπερβολή σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Ε, πολλές φορές ε, ήδη στατιστικά δεδομένα υπάρχουν στις εθνικές υπηρεσίες. Δεν θα, πρέπει, θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις ε, επικαλύψεις και θα πρέπει να φροντίσουμε να λειτουργεί σωστά η συγκέντρωση και η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων. Όσον αφορά τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, θέλουμε να τονίσουμε ότι η συνεργασία με τις εθνικές αρχές είναι σημαντική. Ε, και εδώ υπάρχει δέσμευση της ε, εμπιστευτικότητας. Και πέρα από αυτό θα ήθελα να τονίσω το, την εθνική ε, διάσταση. Επίσης, όσον το θέμα του ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητας όσον αφορά την ε, επιβολή κυρώσεων. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένας διεθνής ε, διάλογος και συνεργασία της ΕΚΤ με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ο κ. Μαυρίδης για Thank you. Ευχαριστώ. Αυτή η αναθεώρηση του πιστάμενου κανονισμού που αφορά τι εξουσίε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την επιβολή κυράσεων σε επιχειρήσει, διότι δεν συμμορφώνονται με του κανονισμού και τι αποφάσει, ελήφθη ούτω ώστε τα καθήκοντα τη ΕΚΤ να ευθυγραμμιστούν με την ενιαία εποπτικό μηχανισμό και το σχετικό κανονισμό. Το πεδίο εφαρμογή των εξουσιών τη ΕΚΤ να επιβάλλει κυρώσει επεκτάθηκε ούτω ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την επιβολή από την ΕΚΤ όλων των διοικητικών κυρώσεων των σχετιζομένων με τις επιδόσεις των εποπτικών καθηκόντων της. Όσον αφορά αυτό, στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων η πρότασή μας στο Συμβούλιο έχει σαν στόχο τη βελτίωση του κειμένου και αυτό σε αρκετά σημεία, συμπεριλαμβανομένων και των κάτω θητριών. Πρώτον, να τονίσουμε ότι η ΕΚΤ θα δρά επί τη βάση ίσης αντιμετωπίσεως των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων άνευ διακρίσεων κατά ιουδήποτε κράτους μέλους. 2. Καθορίζει ότι η περίοδος επιβολής κυρώσεων ξεκινά από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση να ξεκινήσει η διαδικασία κατά παράβαση και όχι η ημερομηνία κατά την οποία διεπράχθη η παράβαση. Τρίτον, να εξασφαλίζεται η διαφάνεια δημοσιεύοντας την απόφαση αμελητή, χωρίς τη δυνατότητα να καθυστερήσει η δημοσίευση μέχρι τρία χρόνια μετά τη λήψη της απόφασης, σε περίπτωση που άμεση δημοσίευση θα υπονόμευε τη σταθερότητα των χρηματοσυντικών αγορών. Όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο, εκφράζουμε ανησυχίες μεγάλες όσον αφορά την τροπολογία του ΕΛΚ, που εισάγει ευρύτερη ε, που προβλέπει ανοιχτή καθυστέρηση σε αυτή την εξαίρεση όσον αφορά τι αποφάσει επιβολή κυρώσεων. Και λέει, μέχρι ότου όλα τα νομικά μέσα εφέσεων έχουν, έχουν εξαντληθεί. Αυτή η διατύπωση είναι σε αντίθεση με την αρχή της διαφάνειας. Πιστεύουμε ένθερμα ότι θα μπορούσε να υπήρχε ένας τρόπος να έχουμε μια ισορροπημένη φράση που θα εξυπηρετεί τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, επόμενος ο κύριος Οζόκ για το ECR. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε ε, και κύριοι, η τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση έχει υποσκάψει την εμπιστοσύνη στον τροπεζικό τομέα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σύστημα εποπτείας και επαρκή διαφάνεια, προκειμένου να μπορέσουμε να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Η ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι ζωτική σημασία, αλλά και πάλι πρέπει να προστατεύσουμε τις ευαίσθητες ή τις απόρριτες πληροφορίες. Συμφωνώ επί της αρχής και με τις δύο εκθέσεις και νομίζω ότι οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ισορροπημένες. Όμως ε, φοβάμαι για τον πολιτικό κίνδυνο που πηγάζει από την ε, μεταφορά τέτοιων σημαντικών εθνικών αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διατάξεις αυτές είναι μέρος ενός ε, ευρύτερου παζλ που έχει να κάνει με την ολοκλήρωση των ε, διάφορων συστημάτων, των κρατών μελών και των οικονομικών συστημάτων και δεν είμαι σκεπτικός. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Νιουχάουζεν για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές και όλους τους άλλους συνεδέλφους που συνεισέφεραν σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δουλειά σας. Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι η ανεπαρκής εποπτεία των τραπεζών έχει, είχε επιπτώσεις στην σταθερότητα της οικονομίας. Τώρα από τον Νοέμβριο έχουμε την Τραπεζική Ένωση και οι σημαντικότερες ε, τράπεζες υπόκειται στον, στην εποπτεία της ΕΚΤ και είναι σημαντικό η ΕΚΤ να μπορεί να δράσει ταχαίως ε, και αποτελεσματικά εφόσον ε, διαπιστώνεται μια παραβίαση των κανόνων. Τα θέματα των δύο εκθέσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Πρόκειται για την αξιολόγηση των εκθέσεων. Και εδώ τρία σημεία είναι σημαντικά. Πρώτον, η ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα, μια σωστή εποπτεία ε, είναι σημαντική. Θα πρέπει να αποκατασταθεί διεθνώς η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη και εντός της Ευρώπης. Επίσης, ε, θα, οι ε, κυρώσει έναντι εκείνων των τραπεζών που δεν τηρούν τους κανόνες θα πρέπει να επιβάλλονται. Επίσης ε, θα πρέπει να αποφύγουμε μια οικονομική αστάθεια. Δηλαδή όταν ε, οι τράπεζες ε, παραβιάζουν κάποιους κανόνες θα πρέπει οι διαδικασίες ε, που κινούνται επί παραβάση θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και συνέχεια θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα. Και ένα τελευταίο σημείο αφορά την ε, βελτίωση της ε, ενημέρωσης. Γι' αυτό στηρίζουμε τις αντίστοιχες τροπολογίες. Ματίας για ένα μισή λεπτό. Ε, ε. Ο κύριος Γκίγκολτ για τους πράσινους για ένα μισή λεπτό. Ναι, συντομία κύριοι συνάδελφοι. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητή Κέιτ Σέιμπορν, συμφωνούμε σε αυτή την έκθεση. Δεν υπήρξαν πολλές Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή συνεργασία. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, καταρχήν στο εξή. Το πρώτο αφορά τα στατιστικά στοιχεία για την κοινή διαριέργεια ελέγχων εκ μέρους της ΕΚΤ. Εδώ το πρόβλημα δεν βρίσκεται τόσο στην νομοθεσία όσο στην ε, εφαρμογή. Και διερωτώ με κατά πόσο είναι σωστό η ΕΚΤ ε, μέχρι τα 50.000 ευρώ να καταρτίζει ένα μητρό και στη συνέχεια να καταγράφονται όλες οι, συνά, οι τραπεζικές συναλλαγές σε αυτό το μητρό και διερωτώ κατά πόσο θα έπρεπε να ισχύει η αρχή της αναλογικότητας. Ο κύριος Μπάλτς ε, ανέφερε τους κινδύνους ενός υπερβάλλοντος ε, ζήλου και τις ενδεχόμενες αλληλοεπικαλύψεις. Ε, τώρα, όσον αφορά τι κυρώσει, και αυτό είναι το πιο επίμαχο σημείο, ε, κατά πόσο θα πρέπει άμεσα να δημοσιοποιούνται, έστω και αν ε, υπάρχει μια νομική ένσταση ε, και ε, βεβαίως ε, όσον αφορά το κράτος δικαίου θα πρέπει, δεν θα πρέπει να δημοσιοποιείται ε, η επιβολή μιας ε, κύρωσης εφόσον υπάρχει το δικαίωμα άσκησης ε, προσφυγής στη δικαιοσύνη. Πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία δεν είναι δυνατόν να δημοσιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία γιατί αυτό αντιβαίνει τελικά στον κανονισμό. Ευχαριστώ ο κύριος Σοφλίν για το EFTD για ένα μισή λεπτό. Στην ε, τελευταία συνέδριση τη ΕΚΟΝ είπα στον κύριο Ντράγκη ότι τον λυπόμουν ε, και το ίδιο ισχύει και τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να κάνει όσε προσαρμογέ ad hoc ε, θέλει σε αρμοδιότητε τη ΕΚΤ, αλλά και πάλι θα έχει μια νομισματική ζώνη που δεν θα έχει τα βελτιστά αποτελέσματα. Οποιοδήποτε αίσθημα εθνική μεταξύ των εθνικών πληθυσμών μόνο τότε θα μπορούσε να δημιουργηθεί ή μια ομαλή ε, νομισματική ζώνη ε, θα χρειαζόταν να αναπτύξετε, να αναπτύξει κανείς αδίστακτες πολιτικές που θα παραβίαζαν ε, την πολιτιστική κουλτούρα. Το αποτέλεσμα είναι να ε, καταργήσετε το ευρώ και να υπάρξουν εθνικά νομίσματα και να μπορούν ε, να υπάρχει λογοδοσία στις εθνικές κυβερνήσεις. Ε, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός να προστατεύει την οικονομική δραστηριότητα στα πιο αδύναμα μέρη. Ίσως ε, κατανοούμε το τι προτείνεται για την ΕΚΤ υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, ε, όμως ε, πρέπει να επιτρέψετε στους λαούς της Ευρώπης να περιορίσουν τις ζημίες τους και πρέπει να στείλετε στη χωματερή το ευρώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρουτσεκ είναι επόμενος. Για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ σχεδόν μεσάνυχτα, πήγε. Και αυτό σημαίνει ότι αυτά τα θέματα δεν μας είναι αδιάφορα. Εστιαζόμαστε επί των λεπτομεριών της λειτουργίας της ΕΚΤ. Ταυτόχρονα η κρίση που φοβόμαστε ε, πηγάζει από αλλού. Πηγάζει από το σύστημα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή η τράπεζα λειτουργεί σαν θεσμός που ελέγχει την, τον εφοδιασμό του ευρώ. Τι σημαίνει αυτό. Ο, την, η υποτίμηση του ευρώ ε, είναι υποφελής για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ταυτόχρονα αυτό σημαίνει απώλειες για όλους τους χρήστες του εν λόγω νομίσματος. Έτσι υποτιμάται το νόμισμα. Οι εθνικές οικονομίες παλιά είχαν δικά τους ε, νομίσματα και μπορούσαν να ελέγχουν τις διακυμάνσεις. Τώρα τροφοδοτούμε αυτό το τεράστιο παράσιτο της Ευρώπης που είναι και η πηγή της κρίσης και δεν μπορούμε να μη βλέπουμε το δάσος λόγω του δέντρου, ε, μπαίνοντα σε λεπτομέρειες. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στα εθνικά νομίσματα, τα παραδοσιακά. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος, ο κύριος Φέρμπερ. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ δεν πρόκειται για το θέμα ευρώ ή όχι, αλλά το θέμα είναι πώς ε, εντός της Τραπεζικής Ένωσης η ΕΚΤ ε, θα είναι σε θέση να πληρεί τις λειτουργίες της. Και για να το κάνει χρειάζεται στατιστικό υλικό και θα πρέπει να είναι σε θέση για εκείνες τις τράπεζες όπου έχει αναλάβει κάποια αποπτικά καθήκοντα να μπορεί να επιβάλλει αντίστοιχες ε, κυρώσεις εάν δεν τηρούνται οι διατάξεις, οι κανόνες. Άρα λοιπόν χαιρετίζουμε ως ε, ΕΛΚ τις δύο αυτές ε, προτάσεις. Θα ήθελα να επικεντρωθώ περισσότερο στο θέμα των κυρώσεων γιατί ε, ασχολήθηκα με το θέμα αυτό στο πλαίσιο πολιτικής μου ομάδας. Εδώ δεν θα πρέπει να υπάρχει το διπλό αξιόπινο. Θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώνει τη διαδικασία και μετά να γίνεται η δημοσίευση Δεύτερον, ε, πού πηγαίνουν τα χρήματα και μου κάνει εντύπωση ότι, μέσω των, ε, ότι, προτείνεται μέσω των ε, χρημάτων αυτό να χρηματοδοτείται η λειτουργία αυτού του, μηχανίσμα, του μηχανισμού. Ε, δηλαδή να χρηματοδοτείται η λειτουργία της επιβολής των διοικητικών ε, κυρώσεων. Τώρα, το πώς θα γίνει ένας διεθνής ε, διάλογος. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διεξαχθεί. Ευχαριστώ. Φερνάντες, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η Τραπεζική Ένωση λειτουργεί ο νέος εποπτικός μηχανισμός ήδη άρχισε τις εργασίες του με επικεφαλή στην ΕΚΤ και σύντομα θα έχουμε και ένα ταμείο εξυγίασης τραπεζών δηλαδή θα είναι μια νέα πρωτοβουλία ελπίζουμε και για την εγγύηση των καταθέσεων όμως δυστυχώς ε, σήμερα έχουμε ένα πολύ μικρό κεφάλαιο έχουμε μόνο 55 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό οι σοσιαλιστές παρουσίασαν μια τροπολογία που έχει ως στόχο τη αντίστοιχα ε, έσοδα, τα έσοδα που αντιστοιχούν στις κυρώσεις να μπορούν να τροφοδοτούν και αυτό το Ταμείο Εξυγίανσης. Θέλουμε πρόσθετα έσοδα για αυτό το Ταμείο γιατί θεωρούμε ότι έχει ελλειπή κονδύλια. Για το λόγο αυτό ζητώ να υπερψηφίσετε την τροπολογία μας σε αυτό το κοινοβούλιο γιατί ενισχύει το σχέδιο της Τραπεζικής Ένωσης και συμβάλλει στο να βγούμε ταχύτερα από τη σημερινή κρίση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Λούκε για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτή την έκθεση δεν έχουμε να κρίνουμε τίποτα εφόσον είμαστε υπέρ της Τραπεζικής Ένωσης. Αν είμαστε υπέρ της Τραπεζικής Ένωσης θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η ΕΚΤ θα αναλάβει αυτή την εποπτική λειτουργία. Αλλά αυτό είναι το καυτό σημείο το, το ερώτημα ε, θα πρέπει ένα θεσμικό όργανο το οποίο μας εφοδιάζει με χρήμα θα πρέπει να έχει και τον εποπτικό, ε, θα πρέπει να έχει την εποπτεία, τη διενέργεια του ελέγχου. Ίσως εδώ πρόκειται για μια σύγκρουση συμφερόντων γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τελικά εφαρμόζει και μία συγκεκριμένη ε, πολιτική με το να φροντίζει για την ε, ρευστότητα. Ένα όργανο το οποίο είναι αρμόδιο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα δεν είναι δυνατόν να ασκεί και αυτό τον έλεγχο. Πρόκειται για μια ε, τεράστια διονγκωμένη αρχή η οποία ε, την οποία δεν θα πρέπει να ανεχθούμε και θα πρέπει να τις προσθέσουμε επιπλέον αρμοδιότητες. Συνάδελφοι, σήμερα έχουμε ένα νέο στάδιο στην ιστορία του ευρώ. Εμείς ε, δίνουμε, έχουμε δώσει νέες αρμοδιότητες ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα έχει ε, συστημικές αρμοδιότητες που δεν είχε πριν. Εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε κάποιες αρμοδιότητες και όλο και περισσότερο μας χώνουν το μαχαίρι στο λαιμό, μας λένε ότι το νόμισμα είναι η... και επομένως η κοινωνία απειλούνται. και οι ευρωσκεπτικιστές ε, μας, ε, μας κατηγορούν μάλλον για ευρωσκεπτικισμού ε, όμως εμείς είμαστε κάτω ευρώ γιατί θεωρούμε ότι πρόκειται για μια κακή πολιτική ιδέα και θεωρούμε ότι οι λαοί είναι το θύμα αυτού του μηχανισμού της ενότητας. Είμαστε ρεαλιστές όταν λέμε ότι αυτό το νόμισμα θα πρέπει να εξαφανιστεί. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Οι τράπεζες πολύ συχνά είναι στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεών μας. Το κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα συχνά. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές για τη δουλειά που έκαναν που είναι πολύ καλή. Συμφωνούμε όλοι ότι παγκόσμια κρίση έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Κάποια κράτη-μέλη βγαίνουν από την κρίση, όμως η κρίση αυτή ήταν συνέπεια εσφαλμένων πράξεων των τραπεζών. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα ε, δεν το διαχειρίστηκαν, δεν το έλεγξαν σωστά. Δεν θέλουμε η ιστορία να επαναληφθεί. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διαφυλάσει τα συμφέροντά μας και τα συμφέροντα όλων των επιχειρήσεων. Ε, τραπεζών, οποιοδήποτε. Αν θέλουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα, χρειαζόμαστε ε, το σωστό, τη σωστή ε, προσέγγιση. Οι κανονισμοί μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα παρέμβασης και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Όμως μεγαλύτερες δικαιοδοσίες απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια. Κάτι που περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στόλογιάν έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να υποστηρίξω τις προτάσεις του Συμβουλίου να αυξηθεί να υπάρξει και εποπτική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να υποπτεύει τις πιο σημαντικές τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εξουσία, χωρίς δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, όταν υπάρξουν παραβιάσεις των κανόνων ή των αποφάσεων της ΕΚΤ ε, και λήψη ε, της εξουσίας συλλογής επαρκών πληροφοριών για να παίξει η ΕΚΤ τον εποπτικό της ρόλο ότι αυτή η προσέγγιση θα ήταν επιβλαβής για την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας εποπτείας και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ήθελα η ΕΚΤ και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτές οι συστάσεις επιφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τη διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς και τη σχέση ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κ. Νίντερμάιερ έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και Λόρδε Χίλ. Πρώτα απ' όλα δράτω με τις ευκαιρίες να συγχαρώ ε, και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που ε, έφεραν σε τέρμα τη διαδικασία της Ταπεζικής Ένωσης την προηγούμενη θητεία. Είναι πολύ καλό για όλους μας και για την Ευρώπη και εύχομαι καλή τύχη στην ΕΚΤ. Η διαδικασία έχει φτάσει σχεδόν στο τέρμα για μας αλλά έχουν μείνει κάποια πράγματα που χρειάζεται να τα επεξεργαστούμε και θα πρέπει να πετύχει το στόχο της συνομοθεσία. Αναφέρεται τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση της βοήθειας σε ρευστό όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, όσον αφορά ε, την έκθεση. Είναι πολύ καλή δουλειά που έκανε η ΕΚΟΝ. Να σχολιάσω τις κυρώσεις. Χρειάζεται ισορροπία μεταξύ διαφάνειας και αποτελεσματικότητας και στεναρότητας. Είναι κάτι πολύ δύσκολο στο χρηματοδοτικό τομέα, διότι πολύ ε, πρώιμη ε, δημοσιοποίηση των πορισμάτων μπορεί να είναι μεγάλο σφάλμα. Οπότε χαιρετίζω το συμβιβασμό της Επιτροπής ΑΚΟΝ για στατιστικά στοιχεία. Ο, πρέπει να πω ότι οι απαιτήσει στατιστικά στοιχεία που επιβάλλουν τις κεντρικές τράπεζες ε, πάντα είναι υπερβολικές θα ζητούσα το ΕΚΤ και το Συμβούλιο να εξετάσουν την χρήση της Τραπεζικής Ενώσεως για τη μείωση του βάρους ε, που ε, έφερουν οι στατιστικές υπηρεσίες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριος Μαλετίτς, ε, για 1,5 λεπτό. Κυρία Μαλετίτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Λόρδε Χίλ. Οι Αυτά που χρειάζονται για αποτελεσματική εποπτεία είναι ε, ποιοτικά δεδομένα και επιβολή κυρώσεων. Ε, όλες αυτές οι εκθέσεις ενδυναμώνουν ε, κάτι τέτοιο και ενδυναμώνουν και την Τραπεζική Ένωση και αυτός είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό συμφωνούμε με τις δύο προτινόμενες εκθέσεις και αυτό διαφάνει στη συζήτηση. Εγώ συμφωνώ η ΕΚΤ να μπορεί να είναι σε θέση, ε, για να μπορεί να είναι σε θέση να ασκήσει το ρόλο πρέπει να έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικά στατιστικά δεδομένα, αλλά το σύστημα πρέπει να είναι σαφές και απλό και να λαμβάνει υπόψη και τις εθνικές διαδικασίες. Όταν μιλάμε για κυρώσεις, θα πρέπει η εποπτεία να συνοδεύεται από μέτρα που να ενθαρρύνουν τις τράπεζες ε, να επιλύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν, που επισημαίνονται. Ε, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι και ο καταμερισμός των οροδιοτήτων μεταξύ της ΑΚΤ και των Εθνικών Τραπεζών. Εγώ νομίζω ότι οι εκθέσεις πάντως πηγαίνουν προς την ορθή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάρας για ένα μισή λεπτό. Αξιότιμα κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Λέμε ναι ε, χωρίς επιφυλάξει την Τραπεζική Ένωση και χαιρόμαστε που και οι δύο εκθέσεις ε, προβλέπουν δύο επιπλέον ε, εργαλεία για την δηλαδή στατιστικά στοιχεία από τη μία και από την άλλη πλευρά το μηχανισμό επιβολής κυρώσεων, ούτως ώστε να μπορεί να αναλάβει αποτελεσματικά τις δραστηριότητε τη εντό της Τραπεζικής Ένωσης. Όσον αφορά τα συστατικά στοιχεία, υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε σχέση με την αναλογικότητα, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί σωστά. Όσον αφορά το μηχανισμό κυρώσεων, εμείς λέμε απερίφραστα ναι, γιατί μια ρύθμιση χωρίς κυρώσεις ε, είναι σαν ε, μια γνάθο χωρίς ε, δόντια. Αλλά δεν θέλουμε διπλές ε, ποινές, γι' αυτό θέλουμε μια διάκριση μεταξύ ε, της επιβολής κυρώσεων και της ε, δημοσιοποίησης η οποία θα πρέπει να γίνεται όταν έχουν εξαντληθεί τα ένδικα μέσα. Γιατί ε, στην περίπτωση αυτή δεν θα είχαμε μόνο ένα διπλό αξιόπινο αλλά θα είχαμε και δυσμανείς επιδράσεις σε εκείνες τις και σε εκείνες τις τράπεζες που δεν ε, πλήγονται άμεσα από τον ε, μηχανισμό κυρώσεων. Ε, αυτές οι εξελίξεις αποτελούν ένα περαιτέρω βήμα για ένα πιο βιώσιμο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο κύριος Κίρτσος έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να υποστηρίξω με την παρέμβασή μου την τροπολογία 4, δηλαδή τη διεθνή παγκόσμια διάσταση των κυρώσεων έχω την εντύπωση ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες που λειτουργούν στις ηνωμένες πολιτείες λειτουργούν κάτω από ένα πιο αυστηρό νομοθετικό διοικητικό πλαίσιο από ότι οι αμερικανικές τράπεζες που λειτουργούν στην ευρωπαϊκή ένωση. αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες άνισου ανταγωνισμού σε μια παγκοσμιοποιημένη τραπεζική αγορά και μπορεί να δημιουργήσει έτσι να προκαλέσει ερεθίσματα στην αμερικανική πλευρά για την επιβολή υπέρογκων προστίμων παρατηρώ διαβάζοντας τον διεθνή τύπο ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. νομίζω πάντως ότι με αυτή την τροπολογία κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. κατά τα άλλα η εικόνα θα έλεγα είναι καλή γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πολιτική απόφαση για τραπεζική ένωση παρατηρούμε ότι είναι πολύ ικανός ο διοικητής της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας παίρνει πρωτοβουλίες αποδεικνύεται δυναμικός και αποτελεσματικός. νομίζω ότι και στο λόρδο χιλ οφείλουμε καλά λόγια γιατί κινείται με χαρακτηριστική άνεση και έτσι ε, αποτελεσματικότητα αλλά και τα στελέχη της οικονομικής επιτροπής που είναι αρμόδιοι για όλους αυτούς τους χειρισμούς απέδειξαν την καλή τους ποιότητα. επομένως είναι ένα θετικό μήνυμα σε μια ευρωπαϊκή ένωση που δοκιμάζεται και αμφισβητείται. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα Περνάμε τώρα στη διαδικασία Κατστιάη. Έχουμε δύο ομιλητές, από ένα λεπτό ο καθένας. Ο κύριος Μαριάς. Θα επανέλθω στο ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων. Διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωρίζουμε ότι είναι καθοριστική στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής και μάλιστα με πάρα πολύ αυξημένες αρμοδιότητες. Ταυτόχρονα πλέον αποκτά και τεράστιες εξουσίες εποπτικού ελέγχου και μάλιστα ελέγχει τις 130 συστημικές τράπεζες οι οποίες έχουν το 81% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα. Όμως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ταυτόχρονα είναι και πιστωτής των κρατών. Έχει αγοράσει ήδη στη δευτερογενή αγορά και μάλιστα με σκόντο τουλάχιστον 217 δισεκατομμύρια ευρώ αξίας κρατικά ομόλογα. ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα είναι και μέλος της τρόικας ενεργώντας και ως δίθεν τεχνικός σύμβουλος. έχουμε μια σύγκρουση συμφερόντων μια υπερενισχυμένη ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα χωρίς το αντίστοιχο πολιτικό αντίβαρο απέναντί της. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιέγκας για ένα λεπτό. Παίρνω το λόγο για να καταγγείλω ε, τον ε, ρόλο της ΕΚΤ ε, στο πλαίσιο της εντολής που της δίνεται από το Καστατικό της. Η ΕΚΤ ουσιαστικά διεύρυνε στα πλαίσια της κρίσης τις αρμοδιότητές της και άρχισε να αγοράζει ε, το ε, δημόσιο χρέος ε, και τώρα φτάνει φτάνουμε στο να μιλάμε και ώστε να μπορέσει να αγοράσει και τοξικούς τίτλους έτσι ώστε να γίνει πραγματική χωματερή. Έχουμε ουσιαστικά συνέπειες σε τομείς πολύ σοβαρούς όπως η παιδεία και η υγεία πώς είναι δυνατόν το ίδιος θεσμός να ε, προβαίνει και σε εποπτεία των τραπεζών και να χαράσει και νομισματική πολιτική. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε όλες αυτές τις αρμοδιότητες της ΕΚΤ χωρίς ένα αντάλλαγμα, ε, χωρίς να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος. Όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που συζητάμε αποτελούν πλήρη ανατροπή τον ε, των Θεσμών απαξιώνουν τους πολίτες ε, και δημιουργούμε εδώ και δημοκρατικό έλλειμμα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ε, έχετε μπλε κάρτα από τον κύριο Γκίκολτ. Δέχεστε. Mr. Giegold, 30 uh, seconds uh, for your question. Δέκα δευτερόλεπτα κύριε το πολύ σύντομα πρέπει να πω ότι πραγματικά έχω μπουχτήσει εδώ. Έχουμε μία συζήτηση για δύο πολύ συγκεκριμένα νομοθετήματα. Ορισμένοι βουλευτές μας είπαν γιατί δεν είναι καλό το ευρώ, κάποιοι άλλοι βουλευτές παραπονιούνται για την Τρόικα, εσείς μας κάνετε γενικές δηλώσεις για την ΕΚΤ. Δεν μπορούμε να έχουμε καλές κοινοβουλευτικές συζητήσεις. Έχαμε όλες αυτές τις συζητήσεις, η Τραπεζική Ένωση, ε, για το ευρώ και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να μείνουμε στο θέμα. Πραγματικά με ενοχλεί αυτό και πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση εδώ ή όχι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά αν θέλετε να απαντήσετε μπορείτε παρακαλώ κύριε Βικάς. Ευχαριστώ. Εγώ είχα και άλλα πράγματα να πω, έτσι λοιπόν σας ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση, γιατί μπορώ να συμπληρώσω. Δεν είναι δυνατόν να ε, έχουμε η ΕΚΤ ε, να αναλαμβάνει μόνο τεχνικά καθήκοντα. Πρόκειται για ένα πολιτικό οργανισμό. Είναι λάθος να τις αποδίδουμε μόνο τεχνοκρατικά καθήκοντα. Εμείς δεν θέλουμε να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Επόμενος, ο Λόρδος Χίλ εκ μέρους της Επιτροπής για δύο λεπτά το πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ε, είναι αργά, αλλά η συζήτηση υπήρξε ενδιαφέρουσα και ο κύριος Γκέγκολτ μας επανέφερε στην τεχνική φύση των θεμάτων τα οποία συζητούμε εδώ και νομίζω ότι δείχνει τη σημασία της φάσης εφαρμογή στην οποία μπαίνουμε στο χώρο αυτό των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ε, τονίζει το ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ε, στην αρχή η Επιτροπή ήδη υιοθέτησε την ε, γνωμοδότηση για, την, ε, για τα στατιστικά στοιχεία και θα πράξει το ίδιο και για το θέμα των κυρώσεων. Ε, υπόθηκε εδώ ότι θα πρέπει τα στοιχεία να είναι εμπιστευτικά, θα πρέπει επίσης να υπάρχει αναλογικότητα, θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των οργανισμών και της ανάγκης άσκησης μιας σωστής εποπτείας. Είμαι ευγνώμων προς την ΕΚΤ, η οποία προετοίμασε τις δύο συστάσεις που θεωρώ ότι δίνουν μια καλή βάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε έχουμε έναν ε, ισχυρό και ε, σωστό από νομική άποψη μηχανισμό επιβολής ε, κυρώσεων και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι στενά με το Κοινοβούλιο, με την ΕΚΤ και το Συμβούλιο ούτε ώστε να έχουμε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα το οποίο θεωρώ επιθυμούν και, τα... και βολευτές εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σιόνιμπορ και τον κύριο Γκουαλτιέρ για τις εκθέσεις τους που μας έδωσαν πλούσια τροφή για σκέψεις και ε, επεσήμεναν ορισμένες, ορισμένους, ε, ορισμένες χρήσιμες λύσεις. Ε, ευχαριστούμε. Οι δύο εισηγητές έχουν ο καθένας δύο λεπτά στη διάθεσή του. Ξεκινάμε με τον κύριο Γκουαλτιέρη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι ούτε καν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσω και τα δύο λεπτά, γιατί νομίζω ότι καταλήγω στο εξή συμπερισμά ό,τι αφορά την έκθεση για τη συλλογή στατικών στοιχείων υπήρχε ευρεία συνένεση, αλλά και συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι εμείς ε, αύριο θα έχουμε μία έγκριση με ευρεία πλειοψηφία και εύχομαι το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις συστάσεις μας και αυτές ε, της Επιτροπής. Βέβαια, καταγράφω ορισμένα πολιτικονομικά προβλήματα επί της άλλης έκθεσης και φυσικά θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα κατάλληλες οι δηλώσεις του Επιτρόπου σε σχέση με τις αφιβολίες που υπάρχουν για την νομική βάση και για την ε, συνέπεια με τον κανονισμό SSM, του υποπτικού μηχανισμού. Έτσι λοιπόν ε, και αύριο στα πλαίσια της ψηφορίας για την έκθεση Σβίμπουρ ε, σας ζητώ να λάβετε υπόψη αυτά τα κρίσιμα σημεία. Σας ευχαριστώ. Next, uh, Επόμενη η κυρία Σουίντεμπορν, η οποία έχει το λόγο για δύο λεπτά. Thank you, Mr. Ευχαριστώ. Υπήρξαν κάποια τεχνικά προβλήματα τέτοια ώρα που είναι. Καλώ του συναδέλφου αύριο να στείλουν ένα χειρό μήνυμα προ το Συμβούλιο ότι χρειάζεται αυξημένη διαφάνεια και δημοσίευση όσον αφορά τι κυρώσει. Καταλαβαίνω, όπω διαφάνει απόψε, ότι εκρεμεί κάποιο θέμα που είναι πολύ επίμαχο. Δηλαδή, κατά πόσο επιτρέπεται έφεση πριν την δημοσιοποίηση και είμαι σίγουρη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβουλεύσει καταλήλω στο Συμβούλιο πώ θα πετυχεί την ισορροπία μεταξύ δημοσιοποίηση των πληροφοριών έναντι του δικαιώματο ε, εφέσεω που έχει με εταιρεία. Θα πρέπει να εξισορροπηθούν οι απαιτήσει τη νομοθεσία για τον ενιαίο αποπτικό μηχανισμό τη εκθέσεω με τι διαδικασίε για αποκάλυψη από τι συγμένε εταιρείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κανονισμό για κατάξη αγορά και τι διάφορε ε, οδηγίε σχετικέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σίγουρη θα βρει μια λύση για όλα αυτά και καλό τα μέλη αύριο να στείλουν ένα έγχειρο μήνυμα για την ανάγκη τη δημοσιοποίηση αύριο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σουίνμπερν. Λοιπόν, η κοινή συζήτηση ολοκληρώθηκε. Η ψηφοφορία επί των εκθέσεων θα λάβει χώρα αύριο. Η επόμενη συνεδρία στη θα χώρα αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, από τις 9 μέχρι τις 2 και το απόγευμα επίσης θα συνεχιστεί και τα πρακτικά